Πρώτο θέμα είναι οι ψηφοφορίες ε, για ε, το, θέμα της κατάστασης στη Σρι Λάγκα. Έχουμε, θέτουμε σε ψηφοφορία το σχέδιο ε, της πρότασης ψηφίσματος της ε, Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς και των Πρασίνων. Την θέτουμε σε ψηφοφορία υπέρ... Ψηφίζουμε. Ε, κατά αποχές απορρίπτεται. Ο κύριος Μεντίνα, έχει διαδικαστικό. Και Παρίσταμε σε αυτή τη συνεδρίαση, αλλά δεν συμμετέχω στην ψηφοφορία. Αυτό είναι η συμφωνία που έχουμε κάνει με την ομάδα των σοσιαλιστών. Το καταγράφουμε αυτό. Εν πάση περιπτώσει είχε σαφή πλειοψηφία η... το αποτέλεσμα. Ήταν με σαφή πλειοψηφία. Τώρα ε, εξετάζουμε την κοινή πρόταση ψηφίσματος τεσσάρων πολιτικών ομάδων ε, για το ίδιο θέμα. Δεν έχω τροπολογίες, αλλά ο κύριος Τάνοκ θέλει να προτείνει προφορική τροπολογία. Στην παράγραφο 2, ε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ζητώ μια αλλαγή τη τελευταία στιγμή στη διατύπωση της προφορική τροπολογίας, αν το επιτρέπετε, διότι τώρα έχουμε ξεκαθαρίσει το πρόβλημα. Το non-fire period δεν είχε κανένα νόημα και γι' αυτό βάλαμε ceasefire, δηλαδή εκεχηρία, κατάπαυση πυρός. Και αυτός ο όρος, ο non-fire, χρησιμοποιείται στο κείμενο της ε, διάσκεψης των συμπροέδρων του Τόκιο. Ζητώ λοιπόν να ακολουθήσουμε την επίσημη διατύπωση του κειμένου. Στην τροπολογία που πρότεινε ο κύριος Τάνοκ, σε αυτή την προσαρμογή στο κείμενο, δεν βλέπω την περίπτωση. Ο κύριος Ματσάκης. Νομίζω ότι και κάτι παρακάτω είναι σημαντικό και πρέπει να μας το πει ο κύριος Τάνοκ. Υπάρχει κι άλλη μια μικρή αλλαγή. Πείτε μας την και αυτή κύριε Τάνοκ πριν ψηφίσουμε. Including the word humanitarian. Humanitarian aid, ανθρωπιστική βοήθεια. Το επίθετο ανθρωπιστική προστίθεται να ξέρουμε τι βοήθεια είναι, αλλά το σημαντικό είναι να πούμε no fire period. Στη δήλωση και του, του Πρόεδρου. Το Τάνοκ. Ψηφίζουμε λοιπόν την ο κύριος Ρωμέβα, που από κίνηση μεγάλη ζωντάνια σήμερα υπάρχει. Κύριε Ρωμέβα, έχετε το λόγο. Κοιτάξτε, υπάρχει κάτι ε, το οποίο δεν το κατα... δεν καταλαβαίνω. Θεωρητικά, αυτό που έχουμε για την προφορική τροπολογία είναι ότι το κείμενο το οποίο θα έπρεπε να υπάρχει θα έπρεπε... είναι το ceasefire και όχι το non-fire. Ε, πρόκειται περί αυτού ή εγώ δεν καταλαβαίνω. Ε, από ό,τι έχω καταλάβει, το κείμενο είναι το ceasefire. Ο, ο κύριος Τάνοκ το έκανε σαφές έκανε, πρότεινε την τελική μορφή της προφορικής του τροπολογίας. Αυτό είναι το οποίο θα τροπολογήσει την παράγραφο. Και ζήτησαν αν υπάρχει αντίδραση, δεν υπήρχε αντίδραση, οπότε ψηφίζουμε την, την, ε, την παράγραφο 2 με την τροπολογία όπως την πρότεινε ο κύριος Τάνοκ. Λοιπόν, ψηφίζουμε υπέρ, κατά, αποχές, Εγκρίνεται η παράγραφος 2 όπως τροπολογήθηκε. Ε, επόμενο θέμα μας είναι η, η παράγραφος ε, στο Ρεσιτάλ Κάπα. Έχει ο κύριος Τάνοκ ακόμη μια προφορική τροπολογία. Κύριε Τάνοκ, σας ακούμε. Να Κύριε Τάνοκ. I've just realized it looks like from από ό,τι κατάλαβα και με βάση τη σειρά εδώ που έχει τυπωθεί, ε, εγώ σας διάβαζα την προφορική τροπολογία στο K και ζητώ συγγνώμη για την ε, σύγχυση. Ενώ τώρα τροποποιούμε την παράγραφο 2. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η σύγχυση. Οπότε, αλλάζουμε κάπως τη σειρά, στην ψηφοφορία και σας ζητώ συγγνώμη. Έχει γραφτεί με τη λάθος σειρά εδώ στον κατάλογό μου διάβαζα την αλλαγή στο εκτιμώντας K και όχι στην παράγραφο 2. Ε, αυτό το οποίο ψηφίζουμε, ε, θα το ψηφίσουμε στη συνέχεια. Σας ζητώ συγγνώμη κύριε Πρόεδρε. Άρα να ξαναπάμε πίσω στην ψηφοφορία, στην τροπολογία 2. Αυτό προτείνω. Κύριε Τάνοκ, θα το κάνουμε αυτό, αλλά πρέπει προσεκτικά να τα παρακολουθούμε. Λοιπόν, ψηφίζουμε την παράγραφο 2. Μπορείτε να πείτε την προφορική τροπολογία, κύριε Τάνοκ, που αναφέρεται στην παράγραφο 2. Και οι συνάδελφοι να ακούν προσεκτικά για να τελειώνουμε. Κύριε Τάνοκ, you have the floor. Okay. Uh, Μάλιστα, για την παράγραφο 2, αυτή που είχαμε δει την περασμένη φορά, θεωρεί ότι η στρατιωτική ε, νίκη ε, ως προς το LTT Στου e, ε, στους τίγρες της Ταμίλ δηλαδή, ε, θα, ε, όπως είναι στον κατάλογο ψηφοφοριών, μέχρι το σημείο που λέει μέχρι να βρεθεί βιώσιμη λύση και ειρήνη. Ωραία. Λοιπόν, υπάρχει αντίδραση στην τροπολογία αυτή, δεν βλέπω, τη θέτουμε σε ψηφοφορία, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται η παράγραφος 2 σωστά τροποποιημένη. Πηγαίνουμε τώρα στο ρεσιτάλ κάπα έχει ήδη τροποποιηθεί και το έχουμε ψηφίσει. Παρακαλώ, κύριε Ματσάκη. Για να τα πούμε σωστά πρέπει να ψηφίσουμε τώρα την ιδεολογική σκέψη K, δηλαδή ΙΑ. Ξαναλέμε την, ε, ε, ιδεολογική σκέψη ΚΑΠΑ. Κύριε Τάνοκ, μπορείτε να ξαναπείτε την, ε, προφορική την προφορική τροπολογία που αναφέρεται σε αυτό το ρεσιτάλ. Θα το πω σωστά για, τον κύριο Ρόμεβα. Καθώς οι ψυμπρόεδροι του Τόκιο ζήτησαν από κοινού, από την κυβέρνηση Σρι και το LTT να δηλώσουν περίοδο no fire για να εκενωθεί η περιοχή από τους άρρωστους και τους ε, πληγωμένους και να παρασχεθεί ανθρωπιστική βοήθεια στον άμαχο πληθυσμό. Πιστεύω δεν υπάρχει τώρα παρεξήγηση. Ψηφίζουμε υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται και το ρεσιτάλ κάπα τροποποιημένο. Τώρα θέτω σε ψηφοφορία το σύνολο της κοινή πρότασης υπέρ, κατά αποχές υπερψηφίζεται. Ε, θα περάσουμε τώρα στην, ε, να δούμε τη σειρά, στην, ψηφο, ψηφοφορία έξι προτάσεων ψηφίσματος σχετικά με την κατάσταση των Βυρμανών προσφύγων στην Ταϊλάνδη ε, ο κύριος Τάνοκ, ε, προτείνει στην παράγραφο 2 μια προφορική τροπολογία. Κύριε Τάνοκ, προσεκτικά η τροπολογία που αναφέρεται στην παράγραφο 2, διότι από ό,τι ξέρω έχετε και για άλλες παραγράφους προφορικές τροπολογίες. Μην τα μπερδέψουμε. Λοιπόν, η τροπολογία ή την παράγραφο 2. Uh, uh, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Βλέπω ότι οι υπεύθυνοι δεν έβαλαν με τη σειρά τις προφορικές τροπολογίες όπως ψηφίστηκαν. Θα είμαι προσεκτική για να βρούμε τη σωστή σειρά. Για την παράγραφο 2 θέλουμε να προσθέσουμε στο τέλος της παραγράφου καθώς και η θελημένη φτώχεια, ε, αυθαίρετη φορολόγηση και ε, δίμευση των κυριών. Ε, βλέπω, λοιπόν, ψηφίζουμε την παράγραφο 2 τώρα, όπως πρότεινε με την τροπολογία του κ. Τάνο, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η τροπολογία και η παράγραφος ψηφίζεται έτσι. Τώρα έχουμε στην ε, παράγραφο 5 στο κείμενο ε, μια επίστροφη προφορική τροπολογία από τον κύριο Τάνοκ. Κύριε Τάνοκ σας ακούμε. Χωρίς μικρόφωνο κύριε Τάνοκ. Ναι, ε, χαιρετίζει τη συνεργασία της κυβέρνησης της Ταϊλάνδης με τον ε, είπα το αρμοστή για τους πρόσφυγες και καλεί και λοιπά για όλους ε, στους ανθρώπους που ζουν στα εισεπλιάρια υπενθυμίζοντας το καθεστώς του πρόσφυγα που θα πρέπει να δοθεί και το πρωτόκολλο σχετικά πρέπει να αναφερθεί. Αρχιαντίθεση. Ψηφίζουμε λοιπόν την παράγραφο με την τροποποίηση αυτή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η τροποποίηση στην ε, παράγραφο 6 τώρα έχετε πάλι προφορική τροπολογία κύριε Τάνοκ σας ακούμε παράγραφος 6 uh, Ευχαριστώ. Θα διαβάσω όλο το κείμενο της 6 όπως τροποποιήθηκε. Υπογραμμίζει ότι οι άνθρωποι που ζουν σε απλία ε, χρησιμοποιούν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η υποστήριξη της κυβέρνησης για να υπάρξει συνεργασία για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό και θα πρέπει ε, αντί για υπουργό να πούμε μόνιμος ε, γραμματέας με τους υπεύθυνους ε, απευθύνει η έκκληση στα μέλη ΑΣΕΑΝ στο Προεδρείο και τους σχετικούς οργανισμούς για να επεξεργαστούν μόνιμη λύση σε αυτό το μακρό πρόβλημα. του κατά αποχές εγκρίνεται άνετα τώρα μετά την παράγραφο 7 έχουμε την τροπολογία των φιλελευθέρων υπέρ κατά ε, κατά είμαστε έτσι αποχές απορρίπτεται ε, έχουμε επίσης την τροπολογία της σοσιαλιστικής ομάδας με ξεχωριστή ε, ψηφοφορία. Το πρώτο μέρος υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Το δεύτερο μέρος θέτουμε σε ψηφοφορία υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τώρα έχουμε μετά την παράγραφο 8 έχουμε ε, τροπολογία των φιλελευθέρων υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και έχουμε τώρα ε, στο, στο ρεσιτάλ ε προφορική τροπολογία. Κοιτάξτε, στο εκτιμώντας ε θα πούμε τα εξής. Ε, ενώ η υπηρεσία προσφύγων των Ηνωμένων Εθνών ανησυχεί για την κατάσταση των προσφύγων και ανησυχεί για την εθνοτική ομάδα των Ροχίνγκια η οποία είναι υποκράτηση από τις Ταϊλανδέζικες αρχές. Υπέρ, ψηφίζουμε υπέρ, το ρεσιτάλ ε, μάλιστα. Ε, κατά, Αποχές. Εγκρίνεται. Και στο, το, θέτουμε το σύνολο σε ψηφοφορία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τώρα ερχόμαστε στο επόμενο θέμα ε, που είναι το κοινό ψήφισμα για το θέμα της έκδοσης του Τσεζάρε Μπατίστη με ε, ονομαστική κλίση. Ανοίγει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Κλείνει η ψηφοφορία. Έχουμε 46 υπέρ και 8 κατά.